Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση για να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας και να ξεκινήσει η τέταρτη ψηφοφορία Επαναλαμβάνεται λοιπόν η συνεδρίαση. Τα αποτελέσματα είναι ως εξής. Ο κανονισμός για την αλλαγή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2017-2020 εγκρίνεται. Συμμετείχαν 479 συνάδελφοι, ψήφισαν 464 υπέρ, 11 κατά και 4 αποχές. Οπότε ο κανονισμός για την αλλαγή του ΠΔΠ εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το δεύτερο τμήμα των τροπολογιών για τα ψηφισμένα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ε, πανδημίας ε, και των αποτελεσμάτων της. Λοιπόν, Υπάρχουν λοιπόν τα αποτελέσματα εκεί πέρα. Στον πίνακα τα βλέπετε, θα δημοσιευτούν και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, τροπολογία 19, όπως βλέπετε, απορρίπτεται ή υπαριθμών 62 τροπολογία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17 Εδάφιο 1 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Εδάφιο 2 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. 3 επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Απορρίπτεται. 64. Απορρίπτεται. 65. Απορρίπτεται.

απορρίπτεται 46 απορρίπτεται 67 απορρίπτεται παράγραφος 20 ε, σε τρία μέρη μέρος πρώτο εγκρίνεται μέρος δεύτερο εγκρίνεται μέρος τρίτο εγκρίνεται τροπολογία 37 απορρίπτεται 68 Απορρίπτεται. 38. Απορρίπτεται. 39. Απορρίπτεται. 40. Απορρίπτεται. 41. Απορρίπτεται. 10. Απορρίπτεται. 23 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Αυτά μέχρι στιγμής ε, για τα αποτελέσματα. Η ψηφοφορία του τρίτου μέρους για το κοινό ψήφισμα για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατοβολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού θα ανακοινωθούν 22 και 50. Περνάμε τώρα στον τέταρτο γύρο ψηφοφορίων. Ψηφίζουμε για το τέταρτο κομμάτι των τροπολογιών για το κοινό ψήφισμα για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανδημία. Η διαδικασία θα γίνει ε, με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινάει η ψηφοφορία από τώρα μέχρι τις 21 και 30. Έχετε μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ ώρα να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή 9 η ώρα το πρωί. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Διακόπτεται η συνεδρίαση. για τόσο λεπτά είναι το Thank you.